τα οποία είναι μη συμβατά με την άσκηση ε, της βουλευτικής τους αρμοδιότητας. Από τις 8 Ιουλίου 2013, σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφο 3 και 4 του κανονισμού, ελέγχθηκαν οι ε, εξουσίες και προτάθηκαν ε, οι θητείες της κυρίας Μπόρζαν, Μπούζικ, Μαλέτιτς, Πετρόβιτς, Γιακοβίνα, Σουίτσα και Τομάζιτς καθώς και των κυρίων Μπαλντίνη, Πίκουλα, Πλένκοβιτς, Στίερ, Βαλγιάλο, Βουλιανίτς. Και αναγνωρίζουμε την έλεξη της θητείας τους κατευθείαν από την 1η Ιουλίου 2013. Οι αρχές της Πολωνίας